πρόεδρο του Συλλόγου Πολωνών της ε, Λευκορωσίας, καθώς και τον κύριο Αλέξανδρο Μιλινκέβιτς, ηγέτη της Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης και βραβευθέντα με το βραβείο Ζαχάροφ το 2006. Ο κύριος Μιλινκέβιτς είναι ηγέτης Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης στην Λευκορωσία και έχει βραβευθεί με το δικό μας βραβείο Ζαχάροφ. Δυστυχώ, ε, η Λευκορωσία ξαναβρέθηκε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων εξαιτία τη δίωξη που ασκήθηκε σε μη κυβερνητικέ οργανώσει. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προασπίζει ανέκαθεν τι οικουμενικέ αξίε ε, τι οποίε ασπάζεται και θα στυλιτεύει τα αυταρχικά καθεστώτα που χρησιμοποιούν την ισχύ του και τη βία και καταδιώκουν δημοκρατικέ οργανώσει μόνο και μόνο επειδή δεν εστερνίζονται τι απόψει του καθεστώτο. Σας έχουν μοιραστεί τα πρακτικά της 11 μέχρι την 11η Φεβρουαρίου.